είστε παρόν στο 50% του χρόνου. Συνεχίζει ο Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λίγη η σημερινή συνεδρίαση. Σας εύχομαι καλό απόγευμα και καλή επιστροφή στα σπίτια σας.